στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Ε, έχω, τα, υπάρχουν ε, νομικές πράξεις που, σχετικά που δημοσιεύονται σε αυτά τα ε, πρακτικά. Η Επιτροπή